εθνική αυτονομία. Με την υπηρεσία αυτή, με την έκθεση αυτό θέλω να επιτύχουμε και σας ευχαριστώ για τις συμβολές σας. So thank you, the Ευχαριστούμε πολύ. Έληξε η συζήτηση. Θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή αύριο στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κάλλας για άλλη μια φορά που ήρθατε εδώ σήμερα. Επόμενο θέμα στην εμερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Ιντουργάη Σαγκούρο που είναι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών για τις διαβουλεύσεις της κατά το έτος 2009. Ο Επίτροπος Σεύτσοβιτς είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Και δίνω το λόγο ευθύ αμέσω στον εισηγητή μας, τον ε, κύριο Ιτουργάη Σαγκούρο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα και μου δίνετε ευκαιρία να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών για το 2009. Οι δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών ε, φέτος, μάλλον πέρυσι το 2009, επηρέστηκε πολύ από το ότι ξεκίνησε η νέα, η 7η κοινοβουλευτική περίοδο. Οπότε άλλαξαν τα μέλη τη Επιτροπή Αναφορών. Τα δύο τρίτα μάλιστα τη Επιτροπή ε, Αναφορών ήταν για πρώτη φορά μέλη τη Επιτροπή Αναφορών. Η έκθεση αυτή προσπαθεί να παρουσιάσει τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2009. Πρώτα απ' όλα να σας εξηγήσω τι σημαίνει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως επίσης και ποιο είναι το αποτέλεσμα της εξέτασης των αναφορών. Η έκθεση αυτή, μάλιστα η ετήσια, εξετάζει και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις συστάσεις που έχουν γίνει παλιότερα για βελτίωση του έργου της Επιτροπής αυτής. Υπογραμμίζει μάλιστα τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η Επιτροπή Αναφορών ε, τώρα που έχει τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας η οποία και επιβεβαίωσε βέβαια το δικαίωμα στην αναφορά για τους Ευρωπαίους πολίτες που αποτελεί θεμελιώδη λίθο των δικαιωμάτων του αλλά ε, προσπαθεί να ενθαρρύνει ακόμα περισσότερο και τους πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Έτσι, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν βελτιώσεις ή να καλυφθούν κενά που υπάρχουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή Αναφορών χαίρεται πάρα πολύ που μπόρεσε να συνεργαστεί βάσει του άρθρου 50 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων προκειμένου να συντάξει έκθεση για την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών που θα είναι έτοιμη στα τέλη της χρονιάς αυτής. Στα ίδια πλαίσια δηλαδή τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να συνεργαστεί περισσότερο με τις αντίστοιχες επιτροπές των Περιφερειακών και Εθνικών Κοινοβουλίων των κρατών μελών με στόχο να υπάρξει ακόμα καλύτερη αμοιβαία κατανόηση όσον αφορά τη διαδικασία των αναφορών και προκειμένου να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν όσο γίνεται πιο γρήγορα ε, απάντηση, ανταπόκριση και λύσει στα προβλήματά του στο καταλληλότερο δυνατόν επίπεδο. Έπειτα ισχύει τώρα, είναι δεσμευτική η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τώρα που άρχισε να ισχύει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Υπογραμμίζει επίση η έκθεσή μα πόσο μεγάλη σημασία έχει η χάρτα αυτή, διότι έτσι γίνονται περισσότερο γνωστά τα δικαιώματα των πολιτών. Πιστεύουμε ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι διαδικασίες προκειμένου να εντοπιστούν όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο καλά τα θεσμικά ζητήματα που έχουν να κάνουν ε, με την Σύμβαση Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που συνυπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζει η Επιτροπή Αναφορών που έχουν να κάνουν ε, με παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησία σε διάφορα κράτη-μέλη. Μα ξέρουμε ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να λύσουν αυτά τα προβλήματα γιατί εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη. Θέλω πάντω να υπογραμμίσω την εξαίρετη συνεργασία που είχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Ιδιαίτερα επίσης να αναφερθώ στις προσπάθειες που έκανε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για να γνωστοποιήσει το έργο του, για να βοηθήσει να λυθούν ε, προβλήματα κακής δίκηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπειτα η προσπάθεια που έγινε για να υπάρξει ένας διοικητικός κώδικας. Εμείς θέλουμε να υπάρξει και ένα διαδικτυακό σύστημα το οποίο να επιτρέπει στον Ευρωπαίο πολίτη να καταλάβει ποια είναι τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, ποιοι είναι οι μηχανισμοί καταγγελίε που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια ενιαία αφαιρίδα για όλα αυτά. Πάντω, θέλω να αποφεληθώ από την ευκαιρία αυτή για να πω ότι από το 2007 υπάρχουν προβλήματα με τις γενικές διευθύνσεις οι οποίες ε, συμπεριλαμβάνουν ε, αναφορές οι οποίες κανονικά δεν είναι σύμφωνες με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι δηλαδή αυτό που εμείς ονομάζουμε ότι δεν είναι αναφορές και που αναγκαζόμαστε όταν τις εξετάζουμε να χάνουμε χρόνο και ανθρώπινους πόρους ε, σε αυτή τη δουλειά χωρίς λόγο, ανθρώπινη ενέργεια. Αυτές είναι 25% ουσιαστικά των αναφορών που λαμβάνουμε. Κάτι τέτοιο όμως η εξέτασή τους, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα αναφορές, ε, κάνει και τους Ευρωπαίους πολίτες να λαμβάνουν περισσότερη καθυστέρηση απάντηση για τα στα προβλήματά τους. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους εκπροσώπους των ε, ευρωπαϊκών ε, ομάδων που συνεργάζονται για να προχωρήσουν οι διαδικασίες στην Επιτροπή Αναφορών. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την Γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών για την βοήθειά της. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ προκειμένου να ετοιμάσουμε αυτή την ετήσια έκθεση τη επιτροπή Αναφορών. Thank you. Can I, can I just ask you... Θα ήθελα ε, αν στο μέλλον χρησιμοποιήσετε τα δύο επιπρόσθετα λεπτά σας να το δηλώσετε εκ των προτέρων. Το λόγο έχει ο Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ιτούρκε για την εξαιρετική του έκθεση και πιστεύω ότι χρειάστηκε πολύ μεγάλη προετοιμασία για αυτή. Νομίζω ότι θα προχωρήσει πέραν αυτών που κατάφερε η κυρία ε, Μαγκίνες, η οποία μας έδωσε, οφείλω να ομολογήσω, μία πλήρη έκθεση. Μετά από τη μελέτη αυτής της έκθεσης βρήκαμε πολλές υποδείξεις για καλύτερη συνεργασία στο μέλλον, διότι θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία των αναφορών αυτών και τον αριθμό τους που ολοένα και διονγκούται. Θα ήθελα επίσης να ε, τονίσω το έργο της κυρίας Ματσόνη, της νέας Προέδρου της Επιτροπής Αναφορών, διότι κατάφερε να δώσει ένα νέο δυναμισμό σε, στις εργασίες αυτής της Επιτροπής. Και υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τις άλλες επιτροπές και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Επιτροπή Αναφορών σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις επιμέρους αναφορές και να βοηθήσουμε εκεί που μπορούμε μελετώντας τα επιμέρους ζητήματα και να έχουμε και μια καλή ανταλλαγή πληροφοριών. Επειδή υπάρχει περιορισμένος χρόνος, θα ήθελα να τονίσω τρία σημεία που είναι άκρος ενδιαφέροντα από πλευράς Κομισιόν. Το θέμα της αναγνώρισης της σημασίας αυτής της συνεργασίας και της συνεργασίας με τα Εθνικά Κοινοβούλια και τις Εθνικές Αρχές. Μίλησε για στενή συνεργασία με τις Επιτροπές Αναφορών στα κράτη-μέλη, διότι πολύ συχνά ό,τι φτάνει στην ευρωπαϊκή, στα ευρωπαϊκά νομοθετικά όργανα προέρχεται από τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, μιλήσατε για φιλικές προς το χρήστη πληροφορίες και ε, επικοινωνία με την Επιτροπή. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι μέσω της διαδικτυακής πύλης θα θέλαμε να ακριβώς εκεί να κατευθύνουμε τους ε, αναφέροντες την τελευταία εβδομάδα φτάσαμε σε μία συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής και το βασικό θέμα ήταν οι διαδικασίες επί παραβάση και βρήκαμε λύση για το θέμα. Ξέρω ότι έχει λήξει ο χρόνος μου, γι' αυτό θα σταματήσω εδώ και αναμένω με προσοχή τη συζήτηση. Έχουμε τώρα τους ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες η κυρία Γκριν εξ ονόματος του ΕΛΚ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να, να συγχαρώ τον συνάδελφο για την έκθεσή του και για το περιεχόμενο του οποίου δεν θα επανέλθω. Θα ήθελα να τονίσω δύο ζητήματα που έθιξε και ο ίδιος ο εισηγητής. Καταρχήν θα πρέπει να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μεταξύ της διαφοράς της ε, πρωτοβουλίας και του ρόλου, που, ε, και του, ρόλου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, τα καθήκοντα που ασκεί. Γιατί στη δική μου εκλογική περιφέρεια βλέπω ότι οι συμπολίτες μου δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη της Επιτροπής Αναφορών. Πώς μπορεί να κινητοποιηθεί καλύτερα λοιπόν ο πολίτης. Χρειάζεται οπωσδήποτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει νέα επικοινωνιακή τακτική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας διαδικτυακός τόπος που να επεξηγεί πώς μπορεί να υποβάλει κανείς μία αναφορά. Επίσης, οι αναφέροντες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της αναφοράς τους δια, του διαδικτύου. Χρειάζεται μεγαλύτερη ορατότητα έτσι ώστε οι πολίτες να ξέρουν ότι βρισκόμαστε πλάι τους, ότι τους ακούμε. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να πληρώσουμε αυτό το επικοινωνιακό χάσμα, γιατί δεν πρόκειται για νομοθετικό έργο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικό. Θα πρέπει η Επιτροπή να ανταποκριθεί σε αυτό το στόχο μέρα με τη μέρα. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών, η κυρία Παλιαδέλη, για ένα λεπτό. Ε, thank you very much, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και ως ε, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών προς τον καλό συνάδελφο κύριο Τουργκάης για την πολύ σημαντική αυτή έκθεση που συνέταξε. Κυρίως επειδή αξιοποιώντας στατιστικά δεδομένα επισημαίνει τον κέριο ρόλο της Επιτροπής Αναφορών στην επαφή των Ευρωπαίων πολιτών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παράλληλα με τον θεσμό του ευρωπαίου διαμεσολαβητή στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του στην ευρωπαϊκή ένωση και τους εκπροσώπους της. από την άποψη αυτή η κομισιόν έχει την υποχρέωση και χαίρομαι ότι ο κ. efovi ήδη το έχει δηλώσει με πρόλαβε να συνεργαστεί με τα μέλη της επιτροπής αναφορών στη μείωση της γραφειοκρατικής λογικής και στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση της επιτροπής σε αιτήματα που διευκολύνουν το έργο της επιτροπής αναφορών στην στην επίσημη και τακτική ενημέρωσή της σχετικά με την πρόοδο στις διαδικασίες επί παραβάση και στη δημιουργία μιας νέας διαδικτυακής πύλης που θα ενημερώνει τους πολίτες για τους διάφορους μηχανισμούς καταγγελίας που είναι στη διάθεσή τους σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης και σε εθνικό επίπεδο. ελπίζω πως η επιτροπή θα ε, αντιμετωπίσει με τη δέουσα προσοχή την έκθεση του κ. Τουργκάης και θα αξιοποιήσει τα συμπεράσματά της με στόχο να επιδιώξει την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Harkin for the Liberals. Η κυρία Χάρκιν από τους ε, φιλελεύθερους για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πλήρη του έκθεση. Εγώ ήμουν αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής για έξι χρόνια και ε, άκουγα πολύ προσεκτικά τους αναφέροντες. Το πρώτο που με ενδιαφέρει είναι ότι οι πολίτες έχουν διαφορετική οπτική γωνία ε, ως προς τα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να μπούμε στη θέση των πολιτών. Θέλουμε μία διαδικασία φιλική προς τον πολίτη, να υπάρχει ένας ε, διάβλος επικοινωνίας, να ακούμε δηλαδή τους αναφέροντες και αυτό να είναι καταλήτης για θετικές αλλαγές. Για πολλούς πολίτες οι αναφορές είναι το τελευταίο στάδιο ενός μεγάλου ταξιδιού όπου έχουν απογοητευτεί ιδιαίτερα. Εμείς θα πρέπει να εξομαλύνουμε αυτό το δρόμο και να μετατρέψουμε την ιστοσελίδα μας σε μία φιλική προς τον πολίτη και μονοαπευθυντική επίσης. Θα πρέπει να υπάρχουν έγκαιρες επεξηγήσεις για το τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Επίσης, το θέμα της, ε, του παραδεκτού ε, ανακύπτει κάθε χρόνο. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε στους αναφέροντες τις επιμέρους αρμοδιότητες. Εάν μία αναφορά δεν είναι παραδεκτή, θα πρέπει αυτό να επεξηγείται στον πολίτη και να του γίνονται υποδείξεις για το τι εναλλακτικά μπορεί να κάνει. Η παράγραφος 17 ε, θα πρέπει να τύχει υποστήριξης διότι πολλές φορές δίνουμε παραπλανητικές πληροφορίες. Δυστυχώς οι μικρές επιχειρήσεις υφίστανται οχλήσεις από τις μεγάλες και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς η νομοθεσία έχει επιπτώσει στη ζωή των πολιτών. Εμείς ως νομοθέτες και η Επιτροπή ως αρχή πρωτοβουλίας θα πρέπει να εισακούμε τον ε, πολίτη έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστούμε την κυρία Χάρκιν και κυρία Αόκεν. Εξωνάντες των πρασίνων για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Τουρκάη για την τόσο σημαντική του έκθεση. Είναι μια έκθεση που περιλαμβάνει πολλές σημαντικές ε, παραγράφους. Πιέζω όμω ο χρόνο, οπότε θα επικεντρωθώ μόνο στις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει. Θέλουμε συγκεκριμένα παραδείγματα αν πιστεύουμε ότι οι πολίτες πρέπει να καταλαβαίνουν περί τίνο πρόκειται. Έτσι λοιπόν εμεί συνεργαστήκαμε με εθνικέ και τοπικέ αρχέ και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν μεγάλες ε, παρεξηγήσεις. Δεν καταλαβαίνω, νομίζω ότι κάνουμε μια αφηρημένη δουλειά και ό,τι καλές προθέσεις και αν έχουμε εμείς ε, προκειμένου να προσπαθήσουμε τη δουλειά μας να την κάνουμε έτσι ώστε να είναι πιο οικία απέναντι στους πολίτες, δεν τα καταφέρνουμε. Γι' αυτό θέλω να φροντίσουμε να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει τον τελευταίο λόγο πάνω από τα εθνικά δικαστήρια. Οι πολίτες ε, όμως έχουν πολλές φορές περιπτώσεις που έχουν περάσει από την εθνική δικαιοσύνη και για οικονομικούς λόγους μερικοί δεν μπορούν να φέρουν τις υποθέσεις τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η τροπολογία 4 για μένα είναι η πιο σημαντική. Εδώ δεν πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφεύγει τις ευθύνε τη Αντίθετα, πρέπει να βρούμε νέους τρόπους ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει το νόμο στι χώρες μέλη και όχι να τι αφήνει να γλιτώνουν. Δεν πρέπει να αφήνουν τα πράγματα στην τύχη τους. Τέλος, όσον αφορά τις διαδικασίες της Επιτροπής μας, και εδώ Πολύ σύντομα θέλω να πω ότι η μέθοδος εργασίας που έχουμε λειτουργεί καλά. Μην ξεχνάμε ότι η εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε και ο κύριος Ζιόμπρο τώρα εκ μέρους των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συμφωνήσω και εγώ με τους άλλους προλαλήσαντες και να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή. Θέλω να τονίσω ότι οι επιτροπές ότι η Επιτροπή μάλλον αναφορών λειτουργεί διαφορετικά όντω από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Υπάρχει μια νέα κατάσταση τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα το Κοινοβούλιο είναι εκείνο που πρέπει να έχει τον ρόλο κλειδί όσον αφορά την ε, πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Η Επιτροπή Αναφορών σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και εκείνη. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στον ρόλο που έπαιξε η Επιτροπή Αναφορών που κατάφερε να λύσει ένα πρόβλημα στη Γερμανία όταν τα γερμανικά δικαστήρια αποφάσισαν ότι οι γονείς παιδιών όταν είναι από διαφορετική υπηκότητα είχαν περιορισμένα δικαιώματα. Να σας μιλήσω τώρα λιγάκι και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Είναι και αυτό ένα θέμα που πολύ απασχόλησε την Επιτροπή Αναφορών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέγερ τώρα εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή εκ μέρους της ομάδας μου. Πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με μια έκθεση με πολλές λεπτομέρειες μετά από τις εντατικές εργασίες το 2009 της Επιτροπής Αναφορών. Οι αναφορές όλο και περισσότερο αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο που έχει στη διάθεσή του Ευρωπαίος πολίτης. Αυξήθηκε ο αριθμός τους, όλες οι αναφορές το 2009 είναι περισσότερες από το 2008. Αυτό δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι που θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να χρησιμοποιήσουν για να λυθούν τα προβλήματά τους, είτε πρόκειται για το περιβάλλον, είτε για τα δικαιώματά τους, είτε για την εσωτερική αγορά. Διαπιστώνουμε ότι έχουμε όλο και περισσότερε. Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία κατά σειρά ε, αριθμού αναφορών. Τώρα ελπίζω να μην κερδίσει βέβαια και η Γερμανία την Ισπανία. Πάντως είμαστε σε ένα, στο Μουντιάλ, Είμαστε λοιπόν ένα μέσο που χρησιμοποιούν οι πολίτε για να υποστηρίξουν τα δικαιώματά του. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω να υπογραμμίσω μερικά πράγματα ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρξει μια απλοποίηση της διαδικασίας αναφορών. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε. Έπειτα θέλω να αναφερθώ και στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν πρόκειται για το περιβάλλον και για τα οικοσυστήματα. Εδώ πρέπει να επιταχύνουμε περισσότερο τις διαδικασίες ώστε η απάντηση που παίρνει ο πολίτης να ε, δίνεται πιο γρήγορα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Όταν φτάνει η επιστολή είναι πολύ αργά. Η ζημιά έχει ήδη γίνει στο περιβάλλον. Οπότε εδώ πρέπει να βρούμε τρόπο να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Επίσης πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να βρούμε μηχανισμούς πιο γρήγορους από τη στιγμή δηλαδή που φτάνει η αναφορά μέχρι να ενημερωθεί ο αναφέρον ότι όντως δικαιώνεται και υπάρχει ζημιά στο περιβάλλον, να μην είναι πολύ αργά. Να πηγαίνει υπόθεση στα δικαστήρια πολύ πιο γρήγορα για να προλαβαίνουμε την καταστροφή. Το 2009 το προσπαθήσαμε. Ήταν μια χρονιά για τη χώρα μου, την Ισπανία, πολύ σημαντική. Η Ισπανία ήταν μία από τις χώρες που έχει περισσότερα προβλήματα όσον αφορά την ε, αύξηση των ε, οικοδομών. Δηλαδή χτίσαμε ανεξέλεκτα. Για άλλη μια φορά στο λιμάνι του Γραναβία, πρόσφατα στην Ουέλβα, το είδαμε με την ρήπανση του ποταμού εκεί. Άρα λοιπόν οι αναφορές όσον αφορά το περιβάλλον είναι ένα μέσον αρκετά αποτελεσματικό που έχουμε στη διάθεσή μας, αρκεί να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Είπαμε, όταν υπάρχουν προβλήματα με το περιβάλλον, οι πολίτε πρέπει να βλέπουν πολύ γρήγορα να προχωράει η διαδικασία για να έχουν μια απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μέγερ. Τώρα, η Λεβέρτμαν, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, το δικαίωμα αναφορά ε, καθορίζει τη συνθήκη Αβώνα σαν σημαντικό τμήμα των δικαιωμάτων των πολιτών. Χώρε όπω η Γερμανία και η Ισπανία υποβάλλουν τι περισσότερε ε, ε, η χώρα μου η Αυστρία είναι πολύ απέχει από τους πρώτους. Είμαι πεπισμένη ότι μια ευρεία αποδοχή από το κοινό θα έχει σημαντικές ε, επιπτώσεις σε θετική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Μέσω μιας αναφοράς οι πολίτες μπορούν άμεσα να έρθουν σε επαφή με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θεσμικά όργανα που συχνά θεωρούνται πολύ ασαφή και γραφειοκρατικά. Αλλά και τα θεσμικά όργανα θα κερδίσουν από αναφορές γιατί πολλές φορές μέσω των αναφορών ε, φαίνεται ξεκάθαρα ο τρόπος εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Παράδειγμα, αμοιβαία ανεξίως ε, αναγνώριση των επαγγελματικών ε, ε, προσόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει διάφορα προγράμματα κινητικότητας. Για να μπορούν να λειτουργήσουν σωστά θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αμοιβαία αναγνώριση των ε, διπλωμάτων. Ε, οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό είναι σωστό να στρέφονται οι πολίτε σε περίπτωση προβλήματος σε εμά. Σαν μέλο τη επιτροπή Αναφοράς, εγώ προσπαθώ να είναι πιο γνωστή και πιο αποτελεσματική αυτή η Επιτροπή. Εάν ξέρουν περισσότερα για τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούν καλύτερα να ελέγξουν και τις μη αποδεκτές ε, ε αναφορές. Τελευταία αναλύση θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεση που παρουσιάσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Βέρτμαν. Θα θα να δώσω το λόγο στην κυρία Μετσόνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω την παρουσία του Επιτρόπου Σευκόβιτς και του εκπροσώπου του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονώνει την έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας για να προωθήσουμε και, τον, και τη δημοκρατική εκπροσώπηση. Εμείς δεν μπορούμε παρά να επαυξήσουμε και να δεχτούμε την επαύξηση των εξουσιών μας. Πρόκειται για το ευρωπαϊκό όνειρο ε, που προέβλεψαν και οι ιδρυτές της κοινότητας. Η πρόσφατη συνθήκη της Λισαβόνας εντάσσει σε αυτό το στόχο την μείζωνα πολι... ε, ε, ε με τη μείζωνα συμμετοχή των πολιτών. Αυτό είναι το κλειδί για τη συμμετοχή των πολιτών στη ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ορίζουμε και την ατζέντα των εργασιών μας. Με βάση τις ενδείξεις και τις υποδείξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής προβάλλουμε και εμείς το έργο μας. Ο συνάδελφος Ιτουργάιτς μας βοήθησε προς τη σωστή κατεύθυνση έτσι ώστε να προωθήσουμε τη συνεργασία Κομισιών Επιτροπής Αναφορών. Έχουμε προωθήσει τις εσωτερικές διεργασίες, πολύ περισσότερες αναφορές γίνονται παραδεκτές και έχουμε ένα σύστημα εξυγχρονισμού χρήσης του διαδικτύου δηλαδή. Κυρία Ματσόνη, θα πρέπει να σταματήσετε γιατί ε, έχετε υπερβεί το χρόνο σας. Έχετε 15 δευτερόλεπτα να συνοψίσετε. Θα ήθελα να τελειώσω μια ευχή για τον επόμενο χρόνο. Ελπίζω να έχουμε μια πιο επικερδή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δέχομαι τα λόγια του κυρίου Σεφκόβιτς. Ελπίζω τα τρία σημεία που προανέφερε να βρουν απήχηση και ελπίζω η δική μας ε, Επιτροπή να διαδραματίσει τον σημαντικό της ρόλο στο νομοθετικό αυτό έργο. Η κυρία Κίνγκα Γκέντς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Έχουμε μία πολύ καλή εικόνα για το 2009. Δεν ήταν εύκολο έτος, διότι τα μέλη της Επιτροπής άλλαξαν κατά τα δύο τρίτα τους και αυξήθηκε και ο αριθμός των αναφορών. Επίσης προωθήσαμε να μειώσουμε το ε, δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο υπήρχε. Ακριβώς αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα μας καθοδήγησε και γι' αυτό επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα για να κινηθούμε υπέρ των πολιτών. Είχαμε ένα πολύ σημαντικό feedback για να δούμε και να προβάλλουμε την εργασία μας ως προς τις non-petitions ο αριθμός τους έχει αυξηθεί και θα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες πότε πρέπει να αποτανθούν στην Κομισιόν και πότε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι αναφορές πολλές φορές αφορούν το ότι δεν έχουν εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη σωστά οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις ιδιαίτερα σε σχέση με το περιβάλλον ή τις ε, πολιτικές ελευθερίες. Βεβαίως, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη αποτελούν πολύ μεγάλο μέρος των περιπτώσεων, των αναφορών δηλαδή που έχουμε δεχτεί. Χωρίς τη βοήθεια του κυρίου Σεκ Σεύκοβιτς δεν θα μπορούσαμε να ήμασταν τόσο αποτελεσματικοί στην επεξεργασία, στη διεργασία αυτή μελέτης των αναφορών. Εάν δεν ε, δράσουμε γρήγορα, δημιουργούνται επιζήμιες καταστάσεις για τον αναφέροντα. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε μεγαλύτερη ταχύτητα, ιδιαίτερα ως προς τις μεταφράσεις προς όλες τις γλώσσες. Ευχαριστώ κύριε για ένα μισή λεπτό. Το δικαίωμα αναφορά είναι ένα πιο σημαντικά δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι μπορούμε να ε, καταγγείλουν ε, ε, παραβίαση των δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, οι αναφορές που βάλουν είναι μια καλή δυνατότητα καταμέτρησης της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαίου και γι' αυτό χαίρομαι ότι υποβάλλονται Υποβλήθησαν μάλλον το 2009 περισσότερε αναφορέ από το 2008. Από την άλλη μεριά, οι πολίτε έχουν και δικαίωμα μια, σε μια σωστή και γλίγορη απάντηση. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τι διαδικασίε. Καταρχήν, οι λεγόμενε μη αναφορέ δεν θα πρέπει να ε, περνάνε στη, στη συζήτηση φτερών αναφορές για τις οποίες δεν είμαστε υπεύθυνοι θα πρέπει να αποπέμπουν γλίγορα και τέλος θα πρέπει η Επιτροπή Αναφορών να έρχεται περισσότερο σε διάλογο με τον υποβάλλοντα την αναφορά. Οι αναφορές παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και μπορούν έτσι να καταστήσουν την Ένωση πιο ζωντανή για τους πολίτες. Και ελπίζω από κοινού εμείς η Επιτροπή Αναφορών δηλαδή η Εκτελεστική Επιτροπή και η Αρμόδια Διοίκηση να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες προσεχώς και για άλλη μια φορά ευχαριστώ τον εισηγητή για την τόσο καλή του έκθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μπουζουτήλ, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφό μου για την έκθεσή του που είναι πάρα πολύ καλή, είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί πρόκειται από μια σημαντική επιτροπή, την Επιτροπή Αναφορών που είναι η γέφυρα μεταξύ ημών και των πολιτών μας. Στην Επιτροπή αυτή δεν δίνουμε μόνο τη δυνατότητα στους πολίτες να μας μιλήσουν, να έρθουν σε διάλογο μαζί μας, αλλά φροντίζουμε να εισακουστούν οι πολίτες. Αυτή η Επιτροπή είναι πάρα πολύ σημαντική ακριβώς γιατί εκεί ακούγεται η φωνή των αναφερόντων των πολιτών. Εγώ θέλω να αφαιρεθώ σε μια αναφορά που προετοίμασα το 2008 εξ τα Επιτροπής αυτής όσον αφορά ε, εμπορικά, ε, εμπορικά κατάστοιχα που παρασύρουν τους πολίτες να δημοσιεύσουν ε, διαφήμιση για τις επιχειρήσεις τους χωρίς να καταλαβαίνουν εκ των προτέρων ότι αυτό είναι έναντι ε, αντιτίμου και πέφτουν έτσι στην παγίδα σχολεία, βιβλιοθήκες και άλλοι, όχι μόνο επιχειρήσεις. Ε, έχουμε λοιπόν πολλά θύματα αυτών των ε, καταλόγων και είχα προκαλέσει την Κομισιόν να υποβάλει μια πρόταση για να επιληθεί άπαθη διαπαντός το πρόβλημα. Δεν έχει δοθεί ακόμα η κατάλληλη ε, απάντηση και θα επιμείνω να γίνει αυτό και παρακαλώ την Κομισιό να σημειώσει τι παρατηρήσει μου. Πρώτα, ευχαριστώ. Είμαι σίγουρο ότι ο Επίτροπο σημείωσε αυτά που είπατε. Τελευταία ομιλητή είναι η κυρία Κολάσκα Κουλάσκα-Μομπίνσκα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, η ετήσια αυτή έκθεση δείχνει και με πολλές λεπτομέρειες μάλιστα πόσο σημαντικό όργανο είναι η Επιτροπή Αναφορών. Οι πολίτες μας, εξάλλου, μας ενημερώνουν τακτικά για το ότι τα κράτη-μέλη δεν τηρούν πάντα τον Ευρωπαϊκό Νόμο. Ξέρουν ότι η Επιτροπή Αναφορών συζητάει τέτοια θέματα. Πολλές φορές τα κλείνουμε. Χωρίς να ξέρουμε κατά πόσο τελικά τα κράτη-μέλη έθεσαν σε εφαρμογή τις αποφάσεις μας ή όχι. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας μηχανισμός ελέγχου εκ των για να ξέρουμε κατά πόσο τα συμπεράσματά μας έχουν ληφθεί υπόψη ή όχι από τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν είναι καλό, γιατί τι συμπεράσματα να βγάλουμε εμείς μετά αν δεν ξέρουμε κατά πόσο οι συστάσεις μας ελήφθησαν υπόψη ή όχι από τα κράτη-μέλη, καλό θα ήταν να ξέρουμε, να έχουμε ένα feedback για το τι έχει γίνει. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοια αναφορών που έχουν εξεταστεί από την Επιτροπή μας, δεν έχει γίνει τίποτα από ό,τι φαίνεται και μετά ξανάρχονται σε μας οι ίδιες αναφορές. Ένας αναφέρον μας πέστησε την προσοχή για κάτι όσον αφορά την Βαλτική θάλασσα και έναν αγωγό που ετοιμαζόντουσαν να χτίσουν εκεί και που ήταν επικίνδυνος. Το 2006 νομίζω ότι ήρθε αυτή η αναφορά. Εμείς λοιπόν ως Επιτροπή Αναφορών ζητήσαμε να σταματήσουν εκεί τα έργα. Να γίνει πρώτα μια μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου και μετά να δούμε. Μετά τι έγινε. Δεν μάθαμε. Δεν ξέρουμε κατά πόσο έγινε αυτό που έπρεπε ή δεν έγινε και μετά ξανάρθε η αναφορά σε εμά. Ε, λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε οι αναφορέ εκείνε οι οποίε φεύγουν από τα χέρια μα γιατί τι έχουμε κλείσει, τι τύχη τι περιμένει μετά. Πρόεδρο, ωραία, κύριε Μαγκίνε, τώρα για τη διαδικασία Κατσδιάη, για ένα λεπτό. Παρακαλώ, κύριε Μαγκίνε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ ε, τον εισηγητή. Το χρόνο μου θέλω να τον χρησιμοποιήσω για να επιστήσω την προσοχή του σώματος εδώ στην ενημέρωση των εργασιών μας. Έχουμε ξεκινήσει το 2006-2007 ε, που κάναμε μια ερευνητική επιτροπή για την Equitable Life. Και τότε είχαμε μια έκθεση το 2007 που ζητούσε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να αναγνωρίσει τις ευθύνες της και να φροντίσει να αποζημιώσει εκείνους οι οποίοι είχαν ασφάλιστρα από την Equitable Life. Σήμερα πολλοί από εσά μπορεί να συναντήθηκαν με εκπροσώπους των εκλογικών σας περιφερειών που ανησυχούν για την αποζημίωση αυτή. Διότι η αποζημίωση αυτή, από ό,τι φαίνεται, θα καλύψει μόνο το 20%. Όμως η Επιτροπή μας δεν είχε αυτό κατά νου θα ήθελα λοιπόν η Ολομέλειά μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα να το δουν αυτό προσεκτικά και να φροντίσουν η Βρετανική κυβέρνηση να τιμήσει τις υποχρώσεις σας. Το είχε πει η νέα Βρετανική κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν τώρα να μην τηρηθούν οι συμφωνίες και να μην αποζημιωθούν όλοι οι ασφαλιζόμενοι όπως πρέπει. Ευχαριστούμε. Κύριο Αλφάνο τώρα. Παρακαλώ. Θεωρώ ότι η προσφυγή αυτή είναι μία από τις ε, πιο σημαντικές για να μπορέσει ε, ο πολίτης να αποτανθεί στις ευρωπαϊκές αρχές. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα έργο ύψης της σημασίας. Μπορείτε να επιβραδύνετε γιατί δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν, ε, δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν οι διερμηνείς ενδιαφέρομαι για τις αναφορές που ε, υποβλήθηκαν σε σχέση με έργα περιβάλλοντος. Δυστυχώς παρά το άρθρο 5.3 που λέει, που αναφέρει ότι οι βουλευτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα εγγραφά, βλέπω ότι η Τράπεζα Δεδομένων είναι, στην Τράπεζα Δεδομένων έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρθεί αυτή η διάκριση, διότι δεν επιβραβεύει την εργασία της ίδιας της Επιτροπής. Έχουμε λίγο χρόνο, γι' αυτό επιταχύνουμε τους ρυθμούς. Τι να πούμε σε ένα λεπτό. Ναι, αλλά θα πρέπει να γινόσαστε και κατανοητοί, λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Μπασέσκου. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ιτουρκάης για την εργασία του. Η συνθήκη της Λισαβόνας ε, τονίζει το ρόλο των πολιτών οι οποίοι μπορούν να αποτανθούν στις ευρωπαϊκές αρχές. Λοιπόν, ότι αυτές οι αναφορές θα πρέπει να σχετίζονται με ε, δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ζήτησα να υπάρχει ένα διαδραστικό κανάλι επικοινωνίας μέσω ενός διαδικτυακού τόπου. Μόνο έτσι δεν θα υπάρχουν παρεξηγήσεις ως προς τις ε, εθνικές και τις κοινοτικές αρμοδιότητες και θα μειωθεί ο αριθμός των μη παραδεκτών αναφορών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεργαστεί η Επιτροπή με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για τη σύνταξη ειδικών εκθέσεων για να μειωθεί ο αριθμός αναφορών, ιδιαίτερα αυτός που δεν ε, επιβάλλονται. Τα καταφέρατε σε ένα λεπτό. Η κυρία Γιάτεμάκη είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του αυτή που είναι πολύ πλούσια σε πληροφορίες. Εγώ δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Αναφορών, όμως η έκθεση αυτή μου έδωσε μια πάρα πολύ καλή εικόνα για το έργο της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2009. Δείχνει μάλιστα και πόσο χρήσιμη είναι αυτή η Επιτροπή Αναφορών. Οι αναφορές είναι όντως χρήσιμες ακόμα και αν το σύστημα αυτό δεν είναι αρκετά γνωστό στους Ευρωπαίους πολίτες. Να λοιπόν, τι προσπάθειες πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια. Πρέπει οι αναφορές να γίνουν πιο γνωστές, μια που μάλιστα και μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε και την ε, πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή για αυτήν την πρωτοβουλία. Πάντως η Επιτροπή Αναφορών και το έργο της θα μας βοηθήσει να πάρουμε κάποια μαθήματα, να καταλάβουμε και έτσι να φροντίσουμε να ενημερώσουμε σωστά τους πολίτες και να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα αναφορές και ε, πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστούμε. Ο κύριος... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω, λέει ο κύριος Ξύπ, ότι η Επιτροπή Αναφορών ιδιαίτερα στην προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγινε ιδιαίτερα γνωστή εξαιτία κάποιων αναφορών που εξέτασε. Εγώ εδώ θέλω να αναφερθώ στην πρόσβαση στην ενημέρωση από πλευρά των Ευρωπαίων πολιτών. Και εδώ συμφωνώ και με την κυρία Αγρονή για το ότι πρέπει να γίνει περισσότερο γνωστή η διαδικασία αναφορών και να γίνει πιο ορατό το έργο της και οι δυνατότητες προσφυγής αυτήν που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Οι πολίτες μας πρέπει επίσης να γνωρίζουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Πρέπει επίσης να ξέρουν τι αποφάσεις, τι συμπεράσματα έχει βγάλει η Επιτροπή Αναφορών για τις διάφορες αναφορές που έχει εξετάσει. Για παράδειγμα, όσον αφορά το North Stream, τον αγωγό αυτόν, κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα η Επιτροπή, αλλά δεν έγινε γνωστά στους πολίτες. Οι πολίτες με ρωτούν τι έχει γίνει. Ευχαριστούμε. Επόμενος. Πρώτα απ' όλα, θέλω να υπογραμμίσω λέει ο κύριος το σημαντικό ρόλο της Επιτροπής Αναφορών. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη βοήθεια που προσφέρει στους Ευρωπαίους πολίτες. Για τον ε, κοινοπολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντική για πάρα πολλούς πολίτες που ενδιαφέρονται για τα δικαιώματά τους και που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με αυτά. Θέλω λοιπόν εδώ να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή μας Μεταφορών θα πρέπει να συνεργάζεται καλύτερα με τις διάφορες Επιτροπές Αναφορών των Εθνικών Κοινοβουλίων. Επίσης, η Επιτροπή Αναφορών έχει και έναν ελεγκτικό ρόλο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή η δικιά μας Επιτροπή Αναφορών ελέγχει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Λέω θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπό μας. Ακούσατε τις παρατηρήσεις των συναδέλφων εδώ, οπότε παρακαλώ να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να εστιάσω την προσοχή μου στα πιο σημαντικά στοιχεία των παρεμβάσεων. Νομίζω ότι μπορώ να ομαδοποιήσω τις παρεμβάσεις σε τρεις καλύτερη επικοινωνία, καλύτερη πληροφόρηση. Δεύτερον, συνεργασία Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τρίτον, τα θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία επιπαραβάση. Ως προς την επικοινωνιακή μας τακτική θεωρώ ότι θα πρέπει να διαδίδουμε καλύτερα τις πληροφορίες, να επεξηγούμε στους πολίτες, να τους εξηγούμε ποιες είναι οι πρωτοβουλίες, πώς διαφέρουν από τις αναφορές, ποια είναι τα δικαιώματά τους σε σχέση με την προσφυγή μέσω Ευρωπαίου διαμεσολαβητή. Επίσης δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να συνεργαστούμε για αυτή την πληροφόρηση. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα μέσα επικοινωνίας μέσω της διαδικτυακής πύλης. Όπως σας είπα και στα εισαγωγικά μου σχόλια, αυτός ο ιστότοπος προβάλλεται και προβλήθηκε και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, θα προβληθεί το έργο και στην Επιτροπή Αναφορών και θα θέλαμε δεδομένα και από άλλες επιτροπές. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την διαδικτυακή πύλη, πώς μπορούμε να πληροφορούμε καλύτερα τους πολίτες μας. μετά από την έγκριση της πρωτοβουλίας υπέρ των πολιτών θα μπορέσουμε όλοι να συνεργαστούμε και στον νομοθετικό τομέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών, διότι συνεισέφερε ε, κατά πολύ στην ε, σύνταξη του ECI και στο εγγύς και μεσοπρόθεσμο μέλλον το θέμα θα συζητηθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όταν το ECI τεθεί σε εφαρμογή θα δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το μέσον. Ως προς την συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας είπα ότι η Επιτροπή θέλει να προβληθεί αυτή η στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι το θέμα των αναφορών απασχολεί ιδιαίτερα τους πολίτες. Θα πρέπει να δράσουμε εντάχει, χωρίς καθυστερήσεις. Διαφορετικά απογοητεύονται οι πολίτες. Πολλές φορές δεν είναι εύκολο αυτό γιατί πρέπει να γίνει μια διεξοδική νομική μελέτη. Γι' αυτό χρειάζεται περισσότερος χρόνος, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα εξεύρουμε τρόπους επιτάχυνσης των διαδικασιών. Το τελευταίο θέμα είναι η διαδικασία επιπαραβάση. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το θέμα μας απασχολεί πολύ σοβαρά και αυτό το διαπιστώνετε όταν βλέπετε τις διαδικασίες αυτές, δηλαδή το άνοιγμα της διαδικασίας επί παραβάση. Θα θέλαμε όλα τα κράτη-μέλη να τηρούν το κοινοτικό δίκαιο και όλες τις οδηγίες και χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, ανταλλαγή απόψεων, ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την κακή μεταφορά του κοινοτικού δικαίου και μόνο όταν δεν γίνει κάτι τέτοιο τότε χρησιμοποιούμε την διαδικασία αυτή, δηλαδή προσφεύγουμε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με βάση τη διαδικασία αυτή της παράβασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες επί παραβάση και χαίρομαι διότι τώρα υπάρχει κατανόηση, συνεννόηση μάλλον, με βάση τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Και μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και να επηρεάσετε και τα κράτη-μέλη από την θέση που κατέχετε. Ως προς άλλες λεπτομέρειες θα έχω καταγράψει όλα σας τα αιτήματα και θα τα διαβιβάσω στις αρμόδιες αρχές. Ευχαριστούμε τον ε, Επίτροπο. Ο κύριος ε, Ιτουργκάιφ έχει το λόγο αν θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο εδώ. Υπάρχει ένας κοινός άξονας όλες τις παρεμβάσεις που ακούσαμε και αυτός είναι η μεγάλη σημασία που έχει η Επιτροπή Αναφορών επειδή μπορούν να προσφύγουν σε αυτήν χιλιάδες πολίτες εμπιστευόμενοι την Επιτροπή αυτή και προσπαθώντας να λύσουν τα προβλήματά τους. Προβλήματα πραγματικά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή Αναφορών όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι, είναι εκείνη που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη από όλε τις κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Εκεί μπορούν να παρέμβουν οι πολίτες και πρέπει να τη διαφυλάξουμε, να την προστατεύσουμε και να την βελτιώσουμε εκεί που μπορεί να βελτιωθεί έτσι ώστε και το Κοινοβούλιο και οι αναφέροντες να μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, ζητώντα από τον Επίτροπο να σημειώσει, ξέρω ότι θα το κάνει ο Επίτροπος, γιατί πολλές από τις διαμαρτυρίες των συναδέρφων που ακούσαμε σήμερα είναι σωστές. Έχουν δίκιο στα σχόλιά τους που λένε ότι δεν υπάρχει αρκετέ πληροφορίε, ότι παραλύονται κάποιες διαδικασίες, ότι καθυστερούν. Είναι σωστό. Πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Οι αναφορές οι οποίες έχουν ανοίξει παραμένουν ανοιχτές και δεν έχουν ακόμα ε, λυθεί τα προβλήματα, πρέπει να τα κοιτάξουμε και πρέπει να φροντίσουμε να γίνει προσπάθεια ώστε οι διαδικασίες αυτές να ολοκληρωθούν, να βρεθεί μια λύση στις αναφορές αυτές που παραμένουν σε κρεμότητα μετά από πολύ καιρό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Η συζήτηση αυτή για την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών έληξε και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα, επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι οι παρεμβάσεις ενός λεπτού. Λαμπρινίδης πρώτα, παρακαλώ.